υπάρχουν παρατηρήσεις, τα πρακτικά εγκρίνονται. Θα κάνω κάποιες, ενα, κάποιες συνακτήρες παρατηρήσεις στο ξεκίνημα αυτής της ολομέλειας. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε τον κύριο Αμουναλή Ραχμόν, πρόεδρο του Τατζικιστάν, ο οποίος ε, βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, σε επίσημη επίσκεψη. Συνομίλησα με τον Πρόεδρο πριν από λίγο, αναφερθήκαμε στις διμερείς σχέσεις και βεβαίως μιλήσαμε και για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητες στο Τατζικιστάν. Κυρίες και κύριοι, την 4η Ιουνίου ε, ε, είχαμε το γενέθλιο δύο σημαντικών γεγονότων. Το 1989 στις 4 Ιουνίου οι αρχές ε, της ε, λαϊκής ε, Κίνας σταμάτησαν, έδωσαν ένα τέλος της εξεγέρσεις των φοιτητών στην πλατεία Τιέναν Όλοι θυμόμαστε το γεγονός αυτό. Την ίδια ημέρα πριν από τόσα χρόνια στην Πολωνία για πρώτη φορά ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έλαβαν χώρα ελεύθερες κοινοβουλευτικές εκλογές και τα μέλη της ε, αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ε, κέρδισαν και πήραν σχεδόν όλους τους, όλες τις έδρες. Οι εκπρόσωποι της δημοκρατικής αντιπολίτευσης